Αρχίζουμε με τις ε, παρεμβάσεις ενός λεπτού. Ο κύριος Μέντες Δεβίγου έχει το λόγο. Στις 14 ε, Φεβρουαρίου του 2008 του Αγίου Βαλεντίνου αποφασίστηκε τα intergroups να συνεδριάζουν μόνο την Πέμπτη. Έκτοτε προσπαθήσαμε να επιλύσουμε αυτό το σύνδεμα χωρίς ε, να το καταφέρουμε. Τα intergroup σήμερα θα πρέπει να συνεδριάζουν μια ημερομηνία που δεν ε, είναι καλή για μας. Δεν υπάρχουν ούτε αίθουσες, ούτε διερμηνία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς τι θα γίνει με τα intergroup και πώς θα λειτουργούν. Θα ήθελα η διάσκεψη των Προέδρων να το ξανασκεφτεί και να ακυρώσει την απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου του 2008. Εάν δεν το κάνει, λέω φιλικά ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε στην Ολομέλεια, διότι η Ολομέλεια είναι το κυρίαρχο όργανο. Κυρίλοφ, για ένα λεπτό.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 τους ε, πρόσφυγες από την Βουλγαρική Θράκη. Πρόκειται για 80.000 ε, άτομα. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί πολλές φορές και από τις δύο χώρες ε, και σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μετανάστες, αλλά πολλά ιστορικά δεδομένα και ένα πρωτόκολλο του 1926 είναι, μαρτυρούν ότι πρόκειται για πρόσφυγες. Υπάρχουν λοιπόν τα στοιχεία και τα έγγραφα, αλλά είναι αρκετά κοινικό να ζητάει από τους ίδιους τους ανθρώπους αυτά τα στοιχεία και τα έγγραφα. Η Ευρώπη ζητεί από την Τουρκία να ενισχύσει τον διάλογο με τη Βουλγαρία όσον αφορά το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι θα πρετανεύσει η φρόνηση και η καλή βούληση εξ ονόματος των καλών σχέσεων γειτονία μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στον τομέα γάλακτος δεν υπάρχει συμμετρική κατάσταση μεταξύ αγροτών και δικτύου διανομής. Επίσης, οι τιμές τις οποίες δεν μπορέσαμε να δαμάσουμε οδήγησαν σε μείωση κερδών σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ε, αρχή επιθεώρησης στον τομέα του γάλακτος για να έχουμε καλύτερο έλεγχο του όγκου παραγωγής και των τιμών. Έτσι θα προσδιορίσουμε τις ανάγκες της αγοράς και θα δούμε πώς εξελίσσεται το κόστος παραγωγής γάλακτος συστηματικά. Επίσης θα υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα του τομέα ε, έτσι ώστε να μην, γίνουν, να μην γίνονται παρεμβάσεις και επιδοτήσεις όπως γίνονται. Ο κύριος Κρέιμερ για ένα λεπτό. Την ε, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου αναφέρεται στον Επίτροπο κύριο Σιμ Κάλλας, ο είπε το εξή. Η, διαδρομή μεταξύ Πρατισλάβα και Παρισίων είναι μια σημαντική διαδρομή και η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η διασύνδεση. Ε, στους ετεροδρόμους, Συντονιστής ο συντονιστής αυτού του έργου, ο Πίτερ Μπάλας, είπε ότι η σιδερόδρομη ε, είναι μια εθνική υπόθεση εν ώψη των περιορισμένων κονδυλίων όσον αφορά την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων οι σταθμοί και όλες οι υποδομές ε, διαχειρίζονται από τις ε, τοπικές και δημοτικές αρχές. Θα ήθελα να καλέσω το ΣΥΜ ΚΑΛΑΣ σε ένα ανακοινωθέν τύπου να, να επαναλάβει τις μέχρι τώρα θέσεις της Επιτροπής και να πει ότι ο σταθμός, ο σταθμός στην Στουτγάρδη δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στις Βρυξέλλες η λέξη του σειρμού είναι λιτότητα, λιτότητα και πάλι λιτότητα. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Πιστεύω ότι μιλάμε για συλλογική κλοπή από τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα από τους συνταξιούχους. Γι' αυτό γνωρίσαμε ε, ένα μεγάλο κύμα απεργιών. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία. Αυτή είναι η αρχή. Πόσες άλλες γενικές απεργίες και διαδηλώσεις χρειάζονται έτσι ώστε να αλλάξει στάση το κέντρο λήψη αποφάσεων, δηλαδή οι Βρυξέλλες. Θα ήθελα να προβλεφθούν νέα δίκαια μέτρα, όπως αναμένουμε όλοι. Κύριος Σαλαβράκος, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, από δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο και επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία δεν αμφισβητούνται βέβαια, προκύπτει ότι έχει αυξηθεί ανησυχητικά η είσοδος αλλοδαπών, χωρίς έγγραφα από τα βόρεια σύνορα της ελλάδας. η frontex η οποία με τη δράση της έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τις ροές αλλοδαπών από τα βορειοανατολικά θαλάσσια σύνορα δεν έχει επιδείξει τα ίδια αποτελέσματα στα βόρεια χερσαία σύνορα από όπου εισέρχονται πλέον κατά χιλιάδες οι αλλοδαποί δημιουργώντας νέα ασφυκτική κατάσταση. χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αυξήθηκαν κατά 640% σε ένα χρόνο οι συλλήψεις αλλοδαπών στην παραμεθόριο πόλη της Ορεστιάδας, ενώ στα νησιά μειώθηκαν κατά 80%. Εν των ανωτέρων, κύριε Πρόεδρε, έχω να προτείνω, όπως επιγόντως αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο, πρώτον, η δημιουργία γραφείου Frontex στην πλευρά της Τουρκίας στον Ευρωποταμό δεύτερον καταγγέλλω την τουρκία που χρηματοδοτείται αδρά από την ευρωπαϊκή ένωση για το μεταναστευτικό και δεν σέβεται τις υποχρεώσεις του από το πρωτόκολλο της άγκυρας και τρίτον ζητώ να ελεγχθεί το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης που αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ο κύριος Σεγγέντη, για ένα λεπτό. a mai Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να φερθώ στην οικολογική καταστροφή στην Ουγγαρία από τη Λιματολάσπη. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν ήδη από τις πρώτες μέρες τόσο τα θύματα όσο και όλους όσους ε, ε, πλήγησαν. Σημαντικό εδώ είναι να διαπιστώσουμε ότι υπήρξαν μεν πολλά θύματα και η καταστροφή αυτή θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά καλείται να, να υιοθήσει μέτρα πρόληψης μελλοντικών καταστροφών. Ε, συμβάσεις ε, ιδιωτικοποίησης ε, έγιναν και με τον τρόπο αυτό ανέφερε στην εξουσία μια ολιγαρχία. Και αυτές οι, οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης θα πρέπει τώρα να εξεταστούν, ελεγχθούν προσεκτικά πολλά εργοστάσια ιδιωτικοποιήθηκαν και ε, θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι απατεώνες θα πρέπει να περιοριστούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σφένσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, οι κλιματικές συνθήκες μας πλήττουν όλους, διότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να εξεύρουν τις σωστές περιβαλλοντικές λύσεις, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές από τις μεγάλες βιομηχανίες. διότι αυτή η κατάσταση μας πλήττει όλους. Θα πρέπει να προασπιστούμε το περιβάλλον, αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, όμως υπάρχουν διαφορετικές ε, μορφές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος που είναι ιδιαίτερα υψηλές. Εμείς θα πρέπει να κοινοποιήσουμε την κατάσταση εκπομπών από τις μεγάλες βιομηχανίες, διότι γνωρίζουμε και θανάτους από τις εκπομπές αυτές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα σφαιρικά. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Αυτές τις μέρες έγιναν συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια μέσω προμήθειας αερίου από διάφορες ε, πηγές ούτως αν μια νέα κρίση του αερίου στην Ευρώπη. Πρόκειται για την, για μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας και του αγωγού που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα μοντέλο επιτυχίας όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ χωρών. Εάν θέλουμε να το διευρύνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2014, και ε, διεύρυνση των πηγών αερίου θα μας οδηγήσει σε μια φτάρκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν στην περίπτωση αυτή να αλληλοϊποστηριχθούν εφόσον ε, υπάρξει μια νέα κρίση εφοδιασμού με αέριο. Επίσης, οι τιμές του αερίου μπορούν να διαμορφωθούν σε περιφερειακό επίπεδο και δεν θα υπάρχει αποκλειστικότητα ενός μόνο προμηθευτού. Ελπίζω αυτά τα project για την ε, θα οδηγήσουν στην πρόθεση του... της κατασκευής του Ναμπούκου, αλλά επίσης ενός αγωγού που θα οδηγεί από το Αζερβαϊτζάν μέχρι τη Ρουμανία. Ο κύριος Μίσκι για ένα λεπτό. Θα ήθελα να προσέξτε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την εργασία. Την Πέμπτη φεύγουν όλα, όλοι οι βουλευτέ από το Στρασβούργο γύρω στι 130, στι 1 και 30 με συγχωρείτε. Όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχει ένα ειδικό τρένο και εξηγήστε μου τη λογική που διατηρούμε ψηφοφορίες παραδείγματος χάρη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 4 στις 4 το απόγευμα. Πώς μπορείτε να κρατάτε μία ψηφοφορία όταν ξέρετε ότι 95% των βουλευτών έχουν φύγει. Βεβαίω, κανείς δεν θα ακούσει την ομιλία μου, δεν θα δώσετε σημασία και είναι λυπηρό. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, παραβιάζεται η δημοκρατία από την καθεστική τάξη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόεδρος της Βουλής της Ρουμανίας έκανε λανθασμένη καταμέτρηση επίτηδες έτσι ώστε να κερδίσει μία ψηφοφορία και να περάσει ένας νόμος. Αυτό που έχει ε, σημασία λοιπόν είναι να γίνει σωστός υπολογισμός, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι μειώθηκαν οι συντάξεις στη Ρουμανία κατά 25% και έγινε καταμέτρηση συμπεριλαμβάνοντας ένα μέλος, ένα βουλευτή, ο οποίος δεν παρευρίσκεται στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή. Ε, εάν γίνει επανακαταμέτρηση, τότε ένας νόμος δεν θα προωθηθεί στη Ρουμανία. Για ένα λεπτό. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, η σουηδική κυβέρνηση έλαβε μία ενημέρωση όσον αφορά ένα δημοσιογράφο που είναι φυλακισμένο στην Ερυθρέα. Σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση, και βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομολογίας του δικαστηρίου είναι καθήκον όλων να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να πετύχουν την ικανοποίηση των ένομων δικαιωμάτων του Ντάβιτ Ιζάκ. Η Ερυθρέα εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση σε συνάρτηση με την χρηματοδοτική ενίσχυση. Αύριο εκπρόσωποι θα έρθουν να δώσουν την νομική γνωμοδότηση αυτή και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ελπίζω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα θα πιέσουν τον πρόεδρο της Ερυθρέας να σώσει τη ζωή του Ντάβιτ Ίσακ. Ε, ένα το Σεπτέμβριο πήγα μια εβδομάδα στο Καζακστάν με μια αντιπροσωπεία της ΓΟΕ. Το Καζακστάν και ο πρόεδρος του έχουν μια δικτατορία ολοκληρωτική θα έλεγα. Πολλές ομάδες που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα συναντήθηκαν μαζί μας. Πρόκειται για ένα τερατώδες καθεστώς με φρικαλαιότητας. Πολλοί φυλακισμένοι που πρόσφατα ε, απελευθερώθηκαν ε, ανέφεραν βασανιστήρια, ξύλο και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ντροπή που το Καζακστάν πήρε την πρόδρια του ΟΑΣΕ για το 2010 και έχουμε και μεγάλες διασκέψεις του ΟΑΣΕ, στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Ο πρόεδρος Ανεπαγιεύ βρίσκεται σε, θα είναι σε επίσημη επίσκεψη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση την άλλη εβδομάδα θα τον υποδεχθεί και ο πρόεδρος Μπούζικ και όλα αυτά επειδή έχουμε τις πετρελαϊκές εταιρείες ε, τις ευρωπαϊκές που έχουν μεγάλα συμφέροντα εκεί όμως πρόκειται για φρικαλαία υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να πάψει αυτό Nelle ultime settimane δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε 30 ε, άτομα που κάνουν ε, απεργία πείνας διότι θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά αυτόν ο αντιτρομοκρατικός νόμος. Όμως οι δύο μεγάλες ε, ομάδες του Κοινοβούλιο δεν ζήτησαν μία ένα ψήφισμα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η απεργία πείνας, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ιδιαίτερα για τους αυτόχθονες. Μιλάμε για την παγκόσμια δήλωση των δικαιωμάτων των λαών. Και του δικαιώματος για την εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη νομοθεσία έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβάλλει στην κυβέρνηση της Χιλής να ακολουθήσει αυτή ακριβώς την νομοθεσία. Ο κύριος Στογιάννοφ, για ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στις επικείμενη, στην επικείμενη συζήτηση στην ε, Τουρκική Βουλή όσον αφορά το δημοψήφισμα στην Βουλγαρική Βουλή όσον αφορά την ε, προσχώρηση της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, μου έκαναν εντύπωση τα όσα είπε ο κύριος Κύριλοφ, ο οποίος επανέλαβε την ομιλία του επικεφαλής της δικής μου πολιτικής ομάδας στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο πριν από δέκα μέρες. Θα ήθελα να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αυτοί οι άνθρωποι που εκδιώχθησαν αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα παιδιά τους γιατί όταν, εάν τα παιδιά έκλεγαν, οι Τούρκοι θα ερχόντουσαν και θα τα σκότωναν. Όσον αφορά τη γενοκτονία των Αρμενίων, αναγνωρίστηκε από την Τουρκία. Ήταν 50.000 ε, ε, Βούλγαροι σκοτώθηκαν και πάρα πολλοί εκδιώχθηκαν από την ε, Τουρκία. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε όχι στην προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε χθε ότι από το 2008 ασκούσαμε πιέσει στην ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα σωστά μέτρα αλλά δεν βγάλαμε το πρόβλημα στον έξω κόσμο γιατί το eurogroup ήταν ανεπίσημο όργανο. η επιτροπή αφήνει να εννοηθεί ότι το ελληνικό έλλειμμα του 2009 θα ξεπεράσει το 15% από 5% που προέβλεπε το μάιο του 2009. αναρωτιέμαι δέκα μονάδες του αεπ πώς μπορούν να περάσουν απαρατήρητες; και όλα αυτά δεν ήταν γνωστά στους υπουργούς οικονομικών όταν αντί για το eurogroup συνεδρίαζαν ως ecofin που είχε τη θεσμική αρμοδιότητα. το πρόβλημα συνεπώς δεν ήταν τόσο η αδυναμία πρόβλεψης όσο η επικράτηση πολιτικών κριτηρίων. οι έλληνες πολίτες όμως ως ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν είχαν το δικαίωμα να γνωρίζουν. χρειαζόμαστε τελικά μεγαλύτερη ανεξαρτησία των αρχών που παρακολουθούν τα δημοσιονομικά κριτήρια και προπαντός δίκαιη και αυτόματη εφαρμογή των κανόνων προς όλους. Ευχαριστώ. Ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έκλεισε με εντάσεις η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας της 6ης Οκτωβρίου και δεν έγινε συνέντευξη τύπου δήθεν για επιμελητιακούς ε, λόγους. Αυτό που έχει σημασία είναι η ισοτιμία του ΟΑΝ που είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό να ανατιμήσει το νόμισμα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο των δασμών μέσα στα πλαίσια της οικονομίας της ε, Κίνας που εντάσσεται στην ε, οικονομία της αγοράς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανατιμήθηκε το Οάν ε, από 2,2 σε γύρω στα, στο 9, το Οάν δηλαδή, σε σχέση με το ευρώ τις σχέσεις μας με την Κίνα βρισκόμαστε σε δυσμενή θέση λόγω της τιμή των πρώτων υλών και της προστατευτικής τους πολιτικής. Άρα είναι αδύνατον να ανταγωνιστούμε ακόμα και αν γίνει ανατίμηση του ευρώ. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σε δύο εβδομάδες. Mr. Rivellini, you make me look unfair to Κύριε Ριβελίνη, μοιάζω να είμαι άδικο με τους άλλους συναδέλφου. που σα άφησα να μιλήσετε περισσότερο από ένα λεπτό. Προσπαθώ να είμαι δίκαιο με όλους. Σας παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι να τηρείτε το χρόνο σας. Ευχαριστώ. Αν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες αποστάσεις στη μεταφορά αγαθών και τη ζήτηση της αγοράς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η κοινοτική αγορά προμηθεύεται πρόβιο κρέας που απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα σε παράλογες τιμές. Η Ρουμανία είναι η πέμπτη χώρα σε παραγωγή πρόβιου κρέατος. Παρόλα αυτά, ε, βλέπουμε ότι οι εξαγωγές μας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Εάν λάβουμε υπόψη ότι μακροχρόνια θα υπάρξουν πολλές οικονομικο-κοινωνικές ε, ταραχές και επειδή μιλάμε για μία προαιώνια παράδοση, θα θέλαμε το Συμβούλιο να μας υποστηρίξει έτσι ώστε να μην αποδυναμωθεί ο τομέας του προβίου κρέατος στη Ρουμανία. Ο κύριος Αρσένης για ένα λεπτό κύριε πρόεδρε το 2008 είχαμε τη μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση. Οι τιμές των δημητριακών εκτοξεύτηκαν οδηγώντας σε πείνα τεράστιους πληθυσμούς κυρίως στην Αφρική. Την ίδια χρονιά είχαμε τη μεγαλύτερη παραγωγή δημητριακών. Ε, γι' αυτό το παράδοξο κατηγορήθηκαν τα βιοκαύσιμα. Τελικά αποδείχτηκε ότι υπεύθυνε ήταν οι χρηματοπιστωτικές εταιρείε που μετά τα παιχνίδια στο Nasdaq και τις φούσκες στην κτηματομεσητική αγορά στράφηκαν προς τα χρέη των κρατών και προς τις, βασικές, τις τιμές των βασικών τροφίμων για να κερδοσκοπήσουν. Αυτά τα παιχνίδια οδηγούν σε εξαθλίωση εκατομμύρια συμπολίτε μας στον κόσμο. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε την ανεξέλεκτη δράση αυτών των εταιριών και απαιτείται σήμερα να μπει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αυτών των εταιριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Φιγκορέιδο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πολέμησης ε, της ε, δουλείας, της σύγχρονης δουλείας. Και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τραγωδία που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι θύματα σύγχρονης δουλείας. Αυτή είναι η πιο ζωφερή πλευρά του καπιταλισμού και της νεοαπικιοκρατίας που επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όταν μιλήσαμε για την ε, Παγκόσμια ημέρα κατά της φτώχειας και σήμερα την Παγκόσμια ημέρα κατά της σύγχρονης δουλείας, ε, όλα αυτά μου φαίνονται λίγο ε, ηρωνικά μέσα στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής των κρατών και τη στιγμή που δεν λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πτυχή και συνοχή για την κοινωνική πρόοδο όπως απαιτούν οι εργαζόμενοι σε όλες τις διαδηλώσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. Ο κύριος για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, 67 χρόνια μετά την καθαίρεση του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνη, στο νότιο Τυρόλο διατηρούνται ακόμα φασιστικά μνημεία τα οποία συντηρούνται για, και για τους κατοίκους εκεί είναι μια καθημερινή ανάμνηση μια αδικοπραγίας. Ε, ο Φράνκο Φρατίνη εδώ και πολλά χρόνια είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός νόμος για την απαγόρευση όλων των ναζιστικών συμβόλων. Νομίζω ότι εδώ εντάσσονται και τέτοιου είδου φασιστικά μνημεία όπως αυτό του Νοτιού Τυρόλου. Νομίζω ότι είναι χρόνος να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτραπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, είναι παραβιάση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει η προστασία των μειονοτήτων να ελέγχεται και να ορίζονται κάποιες ε, συνέπειες σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων αυτών των μειονοτήτων. Yes. Φέτος έχει ανακηρυχθεί έτος κατά της φτώχειας. Ήταν η 23η επέτειο ουσιαστικά του έτους καταπολέμησης φτώχειας, του ΟΗΕ πάντα. Οργανώθηκαν λοιπόν πολλές εκδηλώσεις παγκοσμίω. Ευαισθητοποίηση προς τους αποκλεισμένους από τις κοινωνίες. Η θεωρία είναι ότι θα δείξουμε ε, στο κοινό ότι πρέπει να αντιδράσουμε στην ακραία φτώχεια και ότι είναι προτεραιότητα για όλους μας να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα πρέπει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς τις αιτίε της φτώχειας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων για τους φτωχότερους που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θετική πρωτοβουλία. Όταν μιλάμε για ακραία φτώχεια, πραγματικά η κατάσταση είναι απελπιστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Διεθνής Μέρα κατά της ε, εκμετάλλευσης του ανθρώπου και της σύγχρονης δουλείας θα πρέπει να μας οδηγήσει στο γεγονός θα πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πορνεία προέρχεται από αυτά τα κυκλώματα, γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την ε, αξιοπρέπεια ε, χιλιάδων γυναικών. Γιατί μιλάμε όχι μόνο για το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου, αλλά και την πλέον ε, σύγχρονη μορφή δουλείας. Καταβάλλονται μεγάλες ε, προσπάθειες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γυναίκες είναι τα τελικά θύματα. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι χώρος δράσης. Η επόμενη οδηγία κατά πολέμηση της σύγχρονης δουλείας θα πρέπει να οδηγήσει σε μία μορφή διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν παρόμοια θέματα και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Θα θέλαμε εμείς να είμαστε ο πρόδρομος της αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος. ένα λεπτό. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι εξετάζεται από έναν ανεξάρτητο συμβούλιο που ασχολείται με την αλυσίδα των τροφίμων. Πρόεδρε, δεν είμαι ο μόνος που αναφέρω προβλήματα και η Δανία και η Γαλλία έχουν απαγορεύσει ορισμένες ουσίες που εμφανίζονται στα μπιμπερό των μωρών. Όμως, από την άλλη πλευρά επιτρέπονται για άλλα τρόφιμα Έχουμε και τους ε, τροποποιημένους οργανισμούς που επιτυχαίνουν άδειε. Ο Επίτροπος Δαλή διαφώνησε για το βιφενόλι α την περασμένη εβδομάδα. Ζητώ λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν να γίνει μια ακρόαση της ΕΦΣΑ, της Επιτροπής ε, Γεωργίας και Προστασίας των Καταναλωτών, διότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Πρόκειται για την υγεία τους. Θα ήθελα να από αποτανθώ στον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον Γέρση Μπούζεκ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποστηρίχθηκε το 5 λέ από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο και τα μέτρα λιτότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και λίγες μέρες στην ουσία δεν διαθέτουμε κοινοβούλιο, διότι πέρασε ο νόμος περί συντάξεων με ψευδή καταμέτρηση. Ο κύριος Μπασέσκου ακολουθεί αυτές τις πρακτικές και αυτό σημαίνει και το κόμμα του, το πεντελέ. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πρακτική και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπούζεκ εάν υποστηρίζει το 5L και, το 5 και αν θα υποστηρίζει την κυβέρνηση Μποκ αν παρευρίσκεται σήμερα εδώ. ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε τη λύση στην κρίση. Ορισμένες χώρες τα καταφέρνουν καλύτερα, άλλες έχουν θυγεί βαθύτερα. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ισχυρή αγορά είναι προτεραιότητα και γι' αυτό ανησυχώ από την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει συμφωνία δασμολόγητη με το Πακιστάν. Το Πακιστάν καταλαβαίνω ότι έχει φυσικές καταστροφές, όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία δικαιολογία για να απειλήσουμε το ευρωπαϊκό εμπόριο και ειδικότερα ε, την υφαντουργία. Μιλώ εκ μέρους των εισαγωγών και παραγωγών υφαντουργών της χώρας μου, της Βουλγαρίας. Η χώρα μου είναι μικρή, η κρίση είναι φοβερή και η είσοδος του Πακιστάν στην ευρωπαϊκή αγορά θα απειλήσει την υφαντουργία της Βουλγαρίας. Όταν έχουμε κρίση, Πρόεδρε, Πρέπει να βοηθήσουμε την ε, ε, ευρωπαϊκή αγορά και η είσοδος του Πακιστάν στην αγορά δεν είναι λύση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας επισύρω την ε, προσοχή στην δυσχερή κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η Ρουμανία. Τα μέτρα καταπολέμησης της κρίσης οδηγούν στην καταπολέμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υγεία και στην εκπαίδευση. Έχουμε έναν πληθωρισμό της τάξης του 8%, μείωση του ΑΕΠ και γι' αυτό γνωρίζουμε διαδηλώσεις από όλους τους ε, τομείς, ε, δηλαδή ακόμα και οι αστυνομικοί κατέβηκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Αυτό αφορά και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, εκπαιδευτικούς κλπ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς για να επιτηρήσει την χρηματοπιστωτική πολιτική των κρατών μελών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση που προβάλλει η κυβέρνηση που στην ουσία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Μπαλτσίτης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 10 Οκτωβρίου εξεράγει η πυρκαγιά στο Φέρι Λίσκο Γκλόιερ. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό. Εν πάση περιπτώσει, αποφεύθηκαν ε, θάνατοι, αν θέλετε, αλλά το ατύχημα αυτό κατέδειξε ότι υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια του, ε, των επιβατών. Μετά το, 11 Σεπτεμβρίου ασχοληθήκαμε με την ασφάλεια των επιβατών στα αεροσκάφη. Αφήσαμε όλες όμως τα άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό το ατύχημα κατέδειξε ότι είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε και με τα άλλα μέσα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχα συμμετείχα σε μια αποστολή παρατήρηση των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κυργιστάν και συναντηθήκαμε με πολλούς εκπροσώπους των πολιτικών ε, κομμάτων και του Προέδρου. Ε, και πραγματικά είχαμε την εντύπωση ότι πράγματι η χώρα βρίσκεται στην οδό μετάβασης προς την δημοκρατία παρόλα αυτά υπήρξαν κάποια βία συμβάντα μετά την αποχώρησή μας. Οι ίδιες οι εκλογές διεξήχθηκαν ομαλά. Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι πραγματικά άφλιες. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας και όχι μόνο με το, για το Κυργιζιστάν αλλά και το Τατζικιστάν και το Αφγανιστάν. Είναι υπέρ του κοινού μέλλοντος η εδραίωση της δικής μας παρουσίας στην περιοχή αυτή. Not Και τώρα τελευταίος ομιλητής, αλλά όχι ο λιγότερο σημαντικός, ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε ορισμένα σημαντικά θέματα που έχουμε με την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο. Πρέπει να αποφύγουμε τους κινδύνους του διαδικτύου. Η πρόληψη στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την επιδιόρθωση της σημείας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ασφάλεια στο κυβερνοχώρο. Πρέπει να είναι δυναμική αυτή η ασφάλεια. Πρέπει να προτρέχουμε τον κινδύνο. Η νομοθεσία σε σχέση με το κυβερνοχώρο και το διαδίκτυο δεν πρέπει να περιορίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνολογιών. Χρειαζόμαστε οριζόντια, οριζόντιο συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων ασφάλειας. Χρειαζόμαστε διεθνείς μηχανισμούς συνεργασίας. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιό να επιμείνει όταν έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο. Χρειαζόμαστε μηχο, μηχανισμό για το συντονισμό των εθνικών πολιτικών. Εντάξει είναι η έκθεση του κυρίου Έντβαρτ ε, Κόσουσνικ, το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Τον λόγο έχει ο εισηγητής μας για τέσσερα λεπτά. Eh, Κύριε Πρόεδρε,